Λοιπόν, η ημερησία διάταξη εγκρίνεται. Ας περάσουμε λοιπόν στι ανακοινώσει του Πρόεδρου, στο σημείο 2 της ημερησίας διάταξης. Θέλω να καλωσορίσω τους Ευρωπαίους πολίτες που θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίασή μας, ε, γιατί φυσικά να μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν, ε, από το Τάλιν ε, μέχρι τη Σικελία και από τη Λισαβόνα, στο και Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη δουλειά μας. Σημειώστε το παρακαλώ. Όταν παίρνετε το λόγο να το έχετε κατά νου. Και αν μιλάτε όλοι με σαφήνεια θα είναι και πιο αποτελεσματική και διερμηνία. Η κυρία Λεπέν. Πρέπει να βρίσκεται τώρα ε, στην Γαλλική Εθνοσυλλήψη και η κυρία Λεκπαλιέ θα την αντικαταστήσει εδώ και δεν είναι παρούσα στην αίθουσα. Επίσης, να σας πω ότι στις 28 Ιουνίου η Κορεπέρ κατέληξε σε μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις ε, για την προτιμησιακή μεταχείριση για την Ουκρανία, έτσι ώστε στα τέλη Ιουλίου θα μπορέσει να εγκριθεί αυτό το θέμα οριστικά στο Συμβούλιο. Αυτά για τις ανακοινώσεις. Περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Αν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Και περνάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Πρόκειται για τον εξυγχρονισμό της προστασίας του εμπορίου. Έχει διακοπεί ο τριμερής διάλογος για το θέμα αυτό και τώρα περιμένουμε την νέα όθηση που θα δώσει στον Κυπροεδρία. Στις 12 Ιουλίου την ε, Τετάρτη δηλαδή θα ξεκινήσουμε τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Προεδρία. Για το δεύτερο κεφάλαιο πρόκειται για εναλλακτικές μεθόδους ε, λογιστικής στην ε, περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές τρευλώσεις στην αγορά. Εγώ είμαι αισιόδοξο και πιστεύω θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Εν τέλει, Πολύ γρήγορα έχει καταλήξει σε κοινή θέση το Συμβούλιο. Φυσικά όλα αυτά θα συζητηθούν στον τριμερή διάλογο. Θα έχουμε δύο συναντήσεις περαιτέρω το Σεπτέμβριο στις 20 ε, Ιουνίου αποφασίσαμε τη θέση μας και στις 3 Ιουλίου η Ολομέλεια υπερψήφισε την επανέραξη των τριμερών διαπραγματεύσεων. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Επίσης ε, θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε μια νομοθεσία πριν αποφανθεί ο ΠΟΕ για την υπόθεση Κίνα κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θα μας διευκόλυνε. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να εργαστούμε γρήγορα και περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 4, συγγνώμη 5 της σημερινής διάταξης, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, όλα τα τμήματα. Ο κύριος Μπέγκε ε, είναι εδώ για να μας ε, παρουσιάσει το θέμα. Μπορεί να είμαι πολύ σύντομο σήμερα, απλά να σας ε, υπενθυμίσω ότι είχαμε μια συζήτηση με τον Γενικό εισηγητή Σίκφριντ Μουρεσάν εδώ στην Επιτροπή μας. Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας η Επιτροπή Προπολογισμών του Επιτρόπου Προπολογισμού του Συμβουλίου τοποθετήθηκε στο σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν. Αυτό θα πάει τώρα στην Κορεπέρ. Σήμερα το πρωί μπόρεσα να ρίξω μια ματιά στις λεπτομέρειες ε, που είχαν ε, γίνει. Έχουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε κάθε χρόνο. Λάβαμε τα έγγραφα βέβαια μόλις σήμερα το πρωί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους όχι μόνο να εξετάσουν τις γραπτές προτάσεις ε, για την πρόταση ψηφίσματος, αλλά όταν θα προετοιμάσουν ε, και τις τροπολογίες τους για την τροπολογία για τον προπολογισμό, να δουν επισταμένο στο επίπεδο των πληρωμών και τις προκλήσεις ή τα προβλήματα ή τις επιτυχίες που σημειώνονται για τα διάφορα προγράμματα και στους ε, τομείς που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποια αιτιολόγηση από την ε, Κομισιόν και από το Συμβούλιο αργότερα, γιατί υπάρχουν κάποιες περικοπές, ιδίως ε, στις πληρωμές. Βέβαια, είμαστε στην εξή κατάσταση. Για πρώτη φορά, την τελευταία δεκαετία, κατορθώσαμε να έχουμε μία αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις με τον προπολογισμό για το 2018, βλέπουμε να ξεκινάει η συζήτηση για το πώς θα συζητήσουμε το επόμενο ΠΟΔΙΠ και υπό ποιες προϋποθέσεις. Νομίζω ότι μία από τις ε, καταστάσεις που αντιμετωπίσουμε τώρα εντός του σημερινού πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στις πληρωμές. Δηλαδή, τελειώνουν οι πληρωμές. Έχουμε ένα γενικό νοτοτόριο για τις πληρωμές ε, και για τις ε, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έχουμε συγκεκριμένα νότα όρια σε κάθε κατηγορία. Αυτό κάνει μια διαφορά. Και γνωρίζοντα ότι καταβάλαμε πολλές προσπάθειες για τη μεταναστευτική κρίση και για όλα αυτά τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρχει γενικό πρόβλημα για άλλες προτεραιότητες που σχετίζονται με το εμπόριο και με την κατηγορία της παγκοσμίας Ευρώπης. πριν ε, τις διακοπές, εγώ θα χρησιμοποιήσω το χρόνο που έχω για να θέσω κάποιες ερωτήσεις στην Κομισιόν και να ζητήσω αιτιολόγηση. Αν αιτιολογούνται αυτές οι περιορισμένες περικοπές, όντως. Και πρέπει να δούμε αν θα παρουσιάσουμε και ισχυρή αντίσταση σε σχέση με τα θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Έχουμε την ίδια κατάσταση όπως έγινε και μετά την συμφωνία με τον Ειρηνικό. Και φυσικά ξέρετε ότι είμαι και πρόεδρος ε, της ε, ομάδας για την Κεντρική Αμερική και υπάρχει πραγματική πραγματικό αίτημα να λάβουμε μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν, αυτά ως αρχικά σχόλια για τη συζήτηση. Η πρόταση ψηφίσματος ε, φυσικά βασίζεται σε κάποιους περιορισμούς. Προσπάθησα να επικεντρωθώ σε αυτά τα σημεία, καταρχήν, και κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί η ίδια διαδικασία, γιατί πάντοτε επιμένουμε σε αυτά τα κυρία στοιχεία δηλαδή η κατανομή στην ε, γάμα δέλτα trade να είναι επαρκής έτσι ώστε η Γενική Διεύθυνση να μπορεί να συνεχίσει όλες τις δραστηριότητές της και θα πρέπει φυσικά να, έχουμε, να παρακολουθούμε και το θέμα της ε, διοίκησης, της διαχείρισης. Επίσης, ε, στο πλαίσιο της αναφέρουσης του επόμενου πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να το έχουμε κατά νου Κατόπιν έχουμε το θέμα της διαφάνειας και της εμπλοκής των πολιτών και φυσικά κοινοποίηση των πληροφοριών. Αυτό είναι ένα θέμα που μόνιμα το συζητάμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς τι διαπραγματευόμαστε στους πολίτες, τι κάνουμε και τι ακριβώς παρακολουθεί το Κοινοβούλιο προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο στον εξυγχρονισμό των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Τέταρτον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε στρατηγικές ε, συνεκτικές και για την εξωτερική πολιτική και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πέμπτον, η τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με το εμπόριο και η οικονομική βοήθεια που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία στους εταίρους μας στα ανατολικά σύνορα και στις ε, χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Είναι σημαντικό να συνεισφέρει για τη σταθερότητα σε αυτές τις περιοχές, αλλά και στη Λατινική και Κεντρική Αμερική, αλλά και στην Αφρική. Επίσης, ε, η υψηλότερη χρηματοδότηση της ε, μακροοικονομικής ε, βοήθειας απαιτείται και γίνεται και ένα έτοιμα στην Κομισιό να αξιολογήσει τα εφιστάμενα εργαλεία για την προώθηση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων στη διεθνοποίησή τους σε ό,τι αφορά την συνοχή με άλλα μέσα υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά προς στιγμή και σε ό,τι αφορά τις ε, μεμονωμένες ε, τροπολογίες υπενθυμίζω όσα είπα. Πρέπει να κάνουμε εντατική αξιολόγηση σε σχέση με την ε, αιτιολόγηση των περιορισμένων περικοπών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και φυσικά περιμένω να δω και τις τροπολογίες που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι μέχρι την προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέργκερ. Ο κύριος Σούστα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μόσκορ είναι σκιώδης εισηγήτρια, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και έχει κάποια σχόλια. Θα διαβάζω στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέργκερ για τη δουλειά που έκανε του προπολογισμού. Θέλουμε να κάνουμε ε, τις εκόλουσες παρατηρήσεις. Προτεραιότητες. Η επιστολή για την εντολή που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια τον προηγούμενο μήνα θέτει τις ε, προτεραιότητες, τις οποίες υποστηρίζουμε, όπως την ε, ε, ύπαρξη επαρκών πόρων για το πρόγραμμα και τα προγράμματα ενισχύσεων. Δεύτερον, χωριστές γραμμές προπολογισμού για την ενδιάμεση αξιολόγηση της συμμόρφωσης των τρίτων χωρών. Κατόπιν, η, επένδυση, η στρατηγική ε, για την ανακοίνωση για τη στρατηγική της ε, ε, αποτελεσματικότητας Επαναλαμβάνω ότι έχουμε την, έχουμε, πλήρως υποστηρίζουμε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να υποσημάνω ότι φέτος, αντίθετα με προηγούμενες, προηγούμενες χρονιές, το περιεχόμενο της επιστολής δεν συζητήθηκε με όλες τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζουμε ότι πρόκειται για μια μονομένη περίπτωση και ότι στο μέλλον όλοι θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην έγκριση των προτεραιοτήτων μας. Δεύτερον, η γνωμοδότηση υποστηρίζει είναι υπέρ της ε, άποψης του εισηγητή. Έχουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, ζητάμε και για τη... να δοθούν οι απαραίτητοι πόροι και στην Ανατολική και στην Νότια γειτονία σε αντίστοιχο επίπεδο. Υπό την έννοια αυτή, στην παράγραφο 5 της γνωμοδότησης θεωρούμε ότι ο, όρι, όρος ανατολικό όριο, σύνορο και χώρες που πέρασαν από την ε, Αραβική Άνοιξη μπορεί να είναι παραπλανητική και κάποιες χώρες να μείνουν εκτός του πεδίου. Γι' αυτό θα υποβάλουμε ε, τροπολογία που θα ξεκαθαρίζει τους όρους ε, ανατολική και νότια γειτονία. Επίσης, θέλουμε να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι για να παρακολουθούν τα θέματα του φύλου 4% του, πρωτο, ε, προϋπολογισμού προέρχεται από από τελωνιακούς δεσμούς πρέπει να ε, παραμείνουν οι, βασικοί συγκριτικοί δείκτες όπως έχει συμφωνηθεί για την μέτρηση των επιδόσεων των τελωνιακών διοικήσεων σε επίπεδο κράτους μέλους και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θέλουμε να δοθεί υποστήριξη στην μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να γίνουν μελέτες για τη δημιουργία ενός οργάνου ε, που θα παρακολουθεί το TFA. Τέλος, ένα ταμείο ε, προσαρμογής που θα περικόψει την περιττή γραφειοκρατία η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως γνωρίζετε, η πρόθεση των, του εμπορίου και οι διαπραγματεύσεις ε, για το εμπόριο είναι ε, ε, κατακαιρματισμένες αρμοδιότητες και έχουν και τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ε, αποτέλεσμα σε κάποια στοιχεία των αρμοδιοτήτων Γι' αυτό θα θέλαμε να γίνει μια αναθεώρηση των υφιστάμενων εργαλείων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που θα δημοσιευτούν και θα παρουσιαστούν δημόσια για να, μπορέσει να γίνει καλύτερη κατανόηση των διαφόρων επιπέδων αρμοδιοτήτων. Τέλος, θέλουμε να ζητήσουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένης και της άμυνας να χρηματοδοτείται επιπλέον, από επιπλέον ταμείων και όχι να επιβαρύνει τα υφιστάμενα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ, Μπέντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή, γιατί θεωρώ ότι τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετώπισε έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιπαρερχόμαστε την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί και πιο συγκεκριμένα το σχεδιασμό για τον προπολογισμό και τι πρόκειται να κάνουμε στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού ε, πλαισίου. Προφανώς πρέπει να δούμε πώς θα τα διαρθρώσουμε όλα αυτά στο μέλλον, πώς μπορούν, μπορεί να γίνουν όλα αυτά λειτουργικά, επίσης και σε σχέση με τον Brexit. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Αν κοιτάξετε το σχέδιο γνωμοδότησης εκ μέρους της Επιτροπής. Την προηγούμενη εβδομάδα ως Κοινοβούλιο δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε ε, σε μια κοινή θέση για το έγγραφο εργασία της Κομισιόν προς τα που πηγαίνουμε δηλαδή με συγκεκριμένο περιεχόμενο και όσον αφορά και το εμπόριο. Θα πρέπει για λίγο όσο συζητάμε τη γνωμοδότησή μας να ασχοληθούμε με το πώς ποιες προτεραιότητες θα θέσουμε και πώς θα ε, περιλάβουμε κάποια διορθωτικά στοιχεία στη θέση της Κομισιόν, στο, στο δρόμο που έχει, ξεκινεί, έχει χαράξει η Κομισιόν στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες του εισηγητή οι διάφορες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το εμπόριο και τη χρηματοδότησή του. Για όλα αυτά, με όλα αυτά συμφωνώ. Πρέπει όμως να πω ότι αν δείτε τη σχέση διμερούς και πολυμερούς εμπορίου και στο σχέδιο προπολογισμού θα πρέπει να ενισχύσουμε πιστεύω τον πολυμερή πυλώνα και να εξετάσουμε το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα διάφορα αυτά εργαλεία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, τότε τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να σκεφτούμε πώς εμείς ως Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσουμε την αυτή δομή. Και το επόμενο διήμερο θα συζητά, συζητήσουμε το πολυμερές σκέλος του εμπορικού συστήματος. Και έχω κάποιες ιδέες αν πάμε στο σημείο 4, καταλαβαίνω ποια είναι ακριβώς η προσέγγιση, όμως δεν θα ήθελα να καθορίζεται, να ορίζεται η εμπορική πολιτική ως εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Και η Handelsblatt, ε, ε, η γερμανική εφημερίδα, αναφέρει σε ένα άρθρο ε, για θέματα μεταξύ Υπουργείων. Υπήρχε ένα θέμα αρμοδιοτήτων και δομής. Πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε, να, να, έχω, να ακούσουμε μάλλον τους διάφορους εμπλεκόμενους. Ίσως δεν θα τα καταφέρουμε να το λύσουμε φέτος, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε και να σκεφτούμε την πιθανότητα ενός παρατηρητηρίου εμπορίου, το ένα Trade Watch γιατί αυτό θα διευκολύνει τη διαφάνεια στην εμπορική, της εμπορικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, θα ήθελα όμως να ακούσω την άποψη της Κομισιόν, να ακούσω τι έχουν να πούν για την εισαγωγή ενός τέτοιου μέσου, αν είναι εφικτό να γίνει τώρα ή εν πάση περιπτώσει για το διάστημα 2018-2019. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν γιατί έχουν τεθεί κάποια θέματα. Πρώτον, αναφέρθηκατε το πώς ε, διεκπεραιώνουμε, το πώς ε, τα βγάζουμε πέρα, ε, το muddling through που είπατε στα αγγλικά. Να δούμε τα στοιχεία, τους αριθμούς και πώς θα τεθούν οι προτεραιότητες θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις της Κομισιόν. Αν μπορούν να ε, διευθετηθούν κάποιες από τις εκκρεμίες που μας, η Επιτροπή. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρο και ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά του κυρίου Μπέγκε κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης αλλά και για τις ε, γνωμοδοτήσεις των άλλων ευρωβουλευτών που έχουν διατυπώσει απόψεις. Είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι εν γέννη στηρίζεται τις θέσεις και κυρίως την το εκτεταμένο θεματολόγιο. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, τα την Είναι μια δυσκολία αυτή, όπως επίσης και οι προτεραιότητες, γιατί ε, προωθούμε διάφορες πρωτοβουλίες ταυτόχρονα. Οι βασικές προτεραιότητές μας είναι ξεκάθαρες, αναφέρονται κάθε χρόνο στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και ε, τις τηρούμε, όπως θα δείτε και του χρόνου. Υπάρχει μια ιεράρχηση στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται αυτό φάνηκε και στην ανακοίνωση του εμπορίου για όλους, του Trade for All και θα ενταχθεί και στην ε, ε, αναθεώρηση και στην ε, έκθεση που θα υποβληθεί φέτος και η οποία τώρα συντάσσεται σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση. Εν γέννη θεωρούμε ότι το σχέδιο γνωμοδότησης και ακούγοντας και τις παρατηρήσεις σας ε, μας, μας δείχνουν ότι συμφωνείτε με μάς ότι όλο και περισσότερες, όλο και μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις. Δεν βλέπουμε πάντοτε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά αυτό το παρατηρητήριο του εμπορίου, το Trade Watch. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαπραγμάτευση αλλά και στην υλοποίηση των συμφωνιών μας, να παρακολουθήσουμε την ε, εφαρμογή τους και επ' αυτού συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ελέγχθησαν συμπεριλαμβανομένου και του σκέλους του ε, βιώσιμου εμπορίου. Ο προϋπολογισμός μας είναι σχετικά περιορισμένος, μας επιτρέπει να κάνουμε πολλά κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση, είναι ένας τομέας τον οποίο φυσικά αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Επίσης, υποστηρίζουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνουμε και θέματα ε, εμπορίου και δημοπρατήσεων και επίσης εμπορίου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν τεθεί σχετικά θέματα. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιούμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την πολιτική μας ε, παραδείγματο χάρη κατά την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης και τα γεωγραφικά μέσα, το EMPI ας πούμε, που μας επιτρέπει να ε, υποστηρίξουμε παρκώς ε, την πολιτική γειτονίας και προς και προς Ανατολάς. Αυτή εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για μας και στο θέμα της διαπραγμάτευσης και στο θέμα της υλοποίησης. Όσον αφορά τώρα το Trade Watch, γνωρίζετε τη θέση μας δεν είναι νέα. Σας έχουμε ήδη αναφέρει ότι χρηματοδοτούμε ένα μέρος αυτού του έργου μέσω της χρηματοδότησης του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών. Είναι μια δραστηριότητα που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Κάνουμε τακτικές ενημερώσεις. Η όλη διαδικασία είναι εν εξελίξη, γίνονται όλο και περισσότερες συναντήσεις επί των διαπραγματεύσεων αλλά και των διαφορετικών εμπορικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσει αυτό το έργο. Θεωρούμε ότι με τις δια... Ε, πρωτοβουλίες διαφάνειας που ήδη λειτουργούν συμπεριλαμβανομένων και διάφορων υλικών που υπάρχουν ως ε, κείμενα, έγγραφα διαπραγμάτευσης. Ας πούμε την περασμένη εβδομάδα έγινε η συμφωνία, συμφωνία με την Ιαπωνία που έχει πολιτική υποστήριξη. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη και άρα επαναλαμβάνω απλώς την θέση που ήδη είχαμε διατυπώσει στην Επιτροπή στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέγε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Βεβαίως... Axt haben nehmen müssen, um das eine oder andere rauszunehmen, was man wahrscheinlich ε, όταν ε, κανείς εξετάζει τέτοια κείμενα, είναι απαραίτητο να γίνουν ε, και κάποιες επιλογές, έτσι ώστε αργότερα να μπορούν να προσθεθούν στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν εξ αρχής όλα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Σούστορ για το σημείο 5 και φυσικά με αυτό που είπε ο κύριος Σόλτς όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Είναι, είναι γεγονός ότι τα πλαίσια εντός των οποίων γίνεται η συζήτηση είναι σχεδόν πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής. Ε, εγώ προσπαθώ βέβαια να δω πώς είναι δυνατόν μέχρι τις 14 Ιουλίου να ολοκληρώσω τη διαδικασία γιατί τότε ε, λύγει και η προθεσμία. Ε, α, όχι, 21 του μηνός λύγει η προθεσμία γενικά για τον προπολογισμό, για το κείμενο η προθεσμία για τις τροπολογίες λύγει στις 14 Ιουλίου, ελπίζω να τα καταφέρω. Έχουμε καιρό πάντως και θα έχουμε και χρόνο για να τα συζητήσουμε γιατί η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε ε, Μπέγκε. Σύμφωνα με τις ε, δικές μου πληροφορίες, 21 ε, Ιουλίου λίγη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και ψηφίζουμε στις 30 Αυγούστου. Επομένως, κανένα πρόβλημα, είμαστε απολύτως εντός των χρονικών ορίων. 30 Αυγούστου λοιπόν είναι ε, η σημαντική ε, ψηφοφορία και η σημαντική ημερομηνία. Έχουμε επομένως χρόνο στη διάθεσή μας, κανένα πρόβλημα. Ε, και επομένως ο καθένας μπορεί να υποβάλει ε, τροπολογίες τις οποίες θα έχει καλά σκεφτεί. Πολύ ωραία, ολοκληρώνουμε και το σημείο αυτό. Ε, πριν περάσω στο σημείο 6 θα ήθελα να συγχαρώ τον Κρίστερ Ρόβολτ γιατί είναι πλέον ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ σε αυτήν την Επιτροπή. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6. Τα σημεία 6 και 7 είναι κοινά. Πρόκειται λοιπόν για μια κοινή συζήτηση όσον αφορά την ενισχυμένη, ε, τη Συμφωνία Ενισχυμένη Εταιρική Συμφωνία και Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τη ε, Δημοκρατία του Καζακστάν. Δυστυχώ ο Σλάχο Μπορέλη δεν είναι εδώ. Επομένω θα πω δύο λόγια και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Λοιπόν, ε, η υπογραφή αυτής ε, της ε, ενισχυμένης συνεργασίας έχει ήδη λάβει χώρα από το 2015. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς όμως την ανάμειξη του Κοινοβουλίου, εφήρμοσε την συμφωνία και βεβαίως ε, ήταν μάλλον άτυχη αυτή η διαδικασία γιατί με την Γενική Διεύθυνση Trade είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα υπάρχει έστω και πρόσκαιρη ε, υλοποίηση της συμφωνίας πριν ε, ε, συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο και μάλιστα η ίδια η κυρία Μάλστρομ μας είχε διαβεβαιώσει ότι με αυτόν τον τρόπο ε, θα προχωρήσει η Κομισιόν γιατί άλλωστε είναι και ένα θέμα το οποίο εμείς θέλαμε να αποφασίσουμε σωστά και επομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας. Εν πάση περιπτώσει το Κοινοβούλιο δεν ανεμίχθη καθόλου, το λέω και το ξανατονίζω η νέα συμφωνία ε, δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου ε, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και θα δημιουργήσει επίσης και μια καλύτερη ατμόσφαιρα ε, όσον αφορά τις σχέσεις και με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν να συσφιχθούν ακόμα περισσότερο οι ε, εμπορικέ σχέσει με αυτή τη χώρα. Αρμόδια επί τη ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή ΑΦΕΤ η οποία θα προτείνει ε, σχετική ε, ψηφοφορία, ε, συγγνώμη, σχετική έκθεση όσον αφορά την συμφωνία αυτή. Ο εισηγητής λείπει, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι σήμερα θα πρέπει να γίνει η ανταλλαγή απόψεων και επομένως θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, ίσως να γίνει και μια σύντομη παρουσίαση αυτής της συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης ανάμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καζακστάν. Να πούμε δύο λόγια πρώτα απ' όλα για το Καζακστάν που, βρίσκεται στην, ε, ε, που είναι ε, ο μεγαλύτερος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία και όπως γνωρίζετε αποτελεί και έναν σημαντικό και αξιόπιστο εταίρο όσον αφορά την ενέργεια στην περιοχή. Είμαστε και εμείς, ε, σαν Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, ο πρώτος ε, εταίρος του Καζακστάν. Δεν είναι ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση της χώρας αυτής. Είχαμε επίσης από το 2016 μια εμπορική συμφωνία 21 δις με ένα επιπλέον για το ε, Καζακστάν από τη στιγμή που εισάγουμε ε, ενεργειακούς πόρους. Ε, να σας πω ότι σε όρους αξίας έχει μειωθεί το ποσό λόγω της ανάπτυξης ε, ε, λόγω της αύξησης των προϊόντων. Έχουμε λοιπόν 34 δις ε, για το 2014 και τώρα είμαστε σε 21 δις. Αυτό αφορά όμως την αξία των εμπορικών συναλλαγών και όχι τον όγκο που είναι διαρκής και μπορώ να πω ότι παρουσιάζει και μια αυξητική τάση. Ε, ενισχυμένη λοιπόν συνεργασία με το Καζακστάν. Αυτή είναι η πρώτη ε, ε, συμφωνία νέας γενιάς που, συνάπτονται με τις, που συνάπτουμε με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίω, ε, δεν, αφο... δεν ε, καλύπτονται μονάχα εμπορικά θέματα. Ε, τα εμπορικά είναι το ένα μονάχα πεδίο. Έχουμε άλλα τρία που αφορούν το πολιτικό διάλογο, την συνεργασία σε δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις και επίσης τομεακή συνεργασία. Αυτά είναι τα άλλα τρία πεδία συνεργασία πέραν του εμπορίου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά ε, τη χρονική στιγμή αυτή τη διαπραγμάτευση. Το είπατε κι εσεί άλλωστε στην εισαγωγή σα. Τούτη η συμφωνία ε, από, είχε ολοκληρωθεί όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις το στόχο του 2014 είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2015 τώρα ε, και υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2015 ε, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά από πολλές απόψεις πρώτα απ' όλα Εκείνη την εποχή το Καζακστάν δεν ήταν ακόμα ε, μέλος, μέλος ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Εμπορίου. Και ένα άλλο στοιχείο της χρονικής στιγμής είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα ε, μια στιγμή κατά την οποία ε, οι εντάσεις στην ευρασιατική περιοχή ήταν ε, ιδιαίτερα αυξημένες, αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της Ουκρανίας. Και επομένως η συμφωνία αυτή ε, αποτέλεσε και ένα ισχυρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να εμπλακεί με τις χώρες της ευρωσιατικής οικονομικής σχέσης και επομένως αυτή η Συμφωνία Ενισχυμένης Ειδικής Σχέσης και Συνεργασίας αποτελεί ε, την πρώτη από τις συμφωνίες που συνήθισαν με τις χώρες της ευρωσιατικής Συνεργασίας. Βεβαίως, εντωμεταξύ έχουμε ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις με την Αρμενία και έχουμε ξεκινήσει και διαπραγματεύσουμε με το, με το Κυργιστάν, αλλά ε, το προηγούμενο δημιουργήθηκε με το Καζακστάν. λόγω όλων αυτών ε, των συγκεκριμένων λόγων ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και να αρχίσει να υλοποιείται, να τεθεί ενισχύ. Βεβαίως, τούτη εδώ δεν είναι μια συμφωνία για την οποία η Κομισιόν ή η Γενική Διεύθυνση ε, Trade ε, έχουν ε, τον πρώτο λόγο. Για όλη τη συμφωνία είναι υπεύθυνη η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ωστόσο ε, απεστάλει και επιστολή, κύριε Πρόεδρε, σε εσάς, έτσι ώστε να εξηγηθούν οι ειδικοί λόγοι για τους οποίους σε αυτήν την ε, περίπτωση ε, η υλοποίηση της συμφωνίας και η εφαρμογή άρχισε να υλοποιείται πριν από την πρώτερη συνένεση του Κοινοβουλίου. Επί της ουσίας τώρα, η συμφωνία προ, περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους που στοχεύουν ακριβώς να βελτιώσουν το ε, επιχειρησιακό κλίμα ε, στο ε, Καζακστάν και εν πολλής, σε πολλές περιπτώσεις μάλλον πηγαίνουν πιο πέρα από τα προβλεπόμενα του ΠΟΕ. Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η εξαγωγική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να μειωθεί και το εμπορικό έλλειμμα το δικό μας σε σχέση με το Καζακστάν. Για να σας δώσω ας πούμε ορισμένα παραδείγματα δείγματα ε, για παιδεία για τα οποία ξεπερνάει ε, τα στοιχεία του ΠΟΕ αυτή η συμφωνία. Μπορώ να σας πω τα διανοητικά δικαιώματα. Ε, επίσης η αποφυγή παραλλήλων εισαγωγών ή η καλύτερη, η μεγαλύτερη δέσμευση δέσμη οσον αφορά την σωστή σήμανση των προϊόντων. Επίσης ε, να σας πω ότι έχουμε και στοιχεία ε, διαφάνειας τα οποία κατά πολύ ξεπερνούν τις προβλέψεις του ε, ΠΟΕ και έχουμε και ένα καλό πακέτο για την πρόσβαση στην αγορά για την περιοχή αυτή πέρα και ανεξάρτητα από το γεγονός ε, ότι το Καζακστάν δεν είναι ακόμα ε, πλήρες μέλος της Ευρωσιατικής Συμφωνίας. Επίσης μας δίνει και τη δυνατότητα συμφωνίας ε, στον ενεργειακό τομέα και τον τομέα των πόρων και των ε, υλικών και οπωσδήποτε θα χρησιμοποιηθεί η συμφωνία αυτή έτσι ώστε ε, να ε, ενταχθεί, να εισαχθεί μάλλον και ένα νέο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη. Φυσικά θα, και αυτό είναι η, μεγάλη, η άλλη μεγάλη αγορά, συγγνώμη, διαφορά σε σχέση με, την, με τις προηγούμενες εταιρικές σχέσεις και συμφωνίες τέτοιες είναι ότι πλέον ε, υπάρχει και ε, προνοία σχετικά με την επίλυση διαφωνιών. Τον Μάιο του 2016 λοιπόν τέθησε ισχύ και τον Μάρτιο του 2017 ε, έλεγε χώρα η πρώτη συνάντηση της Εμπορικής Επιτροπής που διέπεται από την συμφωνία αυτή και με χαρά σημειώσαμε στη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης ότι έχει γίνει πρόοδος από πλευράς του Καζακστάν ε, το οποίο έχει λάβει ήδη τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να υλοποιηθούν τα διάφορα πεδία συμφωνίας και οι διάφορες υποχρεώσεις ε, και ε, επίσης είδαμε ότι έχει διευκολυνθεί η κατάσταση όσον αφορά εμπορικά προσκόμματα τα οποία υφίσταντο από πολύ καιρό. Δεν θα πω τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε. Και βεβαίως από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βεβαίως ε, εμείς συστήνουμε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενέσει σε αυτήν την πολύ σημαντική εμπορική συμφωνία. Ευχαριστώ. Είναι έκπληξη αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Παρακαλώ, πρώτος πρώτη σκιώδης. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για τα ευγενικά σας λόγια. Ζητώ συγγνώμη που καθυστόρησα. Δυστυχώς ε, δεν μπόρεσα να ελέγξω τους λόγους καθυστερήσεις που νομίζω με το ίδιο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην ΑΦΕΤ. Είχαμε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καζακστάν. Ανεπίσημα να πω ότι έχω την εντύπωση ότι το Καζακστάν είναι μια σημαντική χώρα σε αυτό το πλαίσιο. Όμως ε, δεν αποτελεί αυτό το κεντρικό σημείο αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Ε, το θέμα είναι η εφαρμογή αυτής ε, της ε, συμφωνίας ε, με έναν εταίρο με τον οποίο έχουμε συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και θα θέλουμε να εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή γιατί έχουν διαρκέσει χρόνια οι διαπραγματεύσεις. Και βλέπουμε το Καζακστάν δεν είναι ακόμα μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, παρόλα αυτά έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διεθνή αρένα σε περιπτώσεις κάποιων σειράξεων, παραδείγματο χάρη στην ε, σύραξη της Συρίας. Πιστεύω λοιπόν ότι υπό το φως των στοιχείων αυτών και αφήνοντα ε, κατά μέρου ε, τα εμπορικά θέματα, θα ήταν καλό να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία σύντομα. Επακόλουθα Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστές διμερείς διαπραγματεύσεις. Η πρότασή μου ίσως είναι να γίνει αυτό σε επίπεδο ΠΟΕ ή τουλάχιστον σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Βεβαίως, πιστεύουμε ότι είναι ζωτικό το Κοινοβουλίο να δώσει τη δική του συγκατάθεση. Αυτό σημαίνει ότι πριν να υπάρξει προσωρινή εφαρμογή πρέπει να γίνει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Αν ε, η Κομισιόν ε, αντιδράσει διαφορετικά, εμείς εκφράζουμε τη λύπη μας. Έχω όμως μία ερώτηση, αν σας κατάλαβα καλά. Νομίζω ότι είπατε ότι έχουμε ένα μηχανισμό για την επίλυση διαφορών. Εγώ δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Ίσως ε, βέβαια αυτό να μην το κατάλαβα καλά γιατί δεν βλέπω να υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Θα ήθελα να με διαφωτίσετε σε αυτό το θέμα. Είναι γενικού τύπου ερώτηση. Και φυσικά υπό το φως της απόφασης ε, της Σιγκαπούρης ε, και σε άλλα πλαίσια σε ό,τι αφορά τη ΣΥΤΑ. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν τι έχει κατά νου. Αλλά θα ήθελα να δω πώς το βλέπει και η Κομισιόν αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, το θέμα αυτό. Πώς βλέπουν αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τους ε, σοσιαλιστές. Είχα κάποιες ερωτήσεις ε, σε σχέση με την κατάσταση με το Καζακστάν που θα έπρεπε να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Καταρχήν, ίσως πρέπει να θέσουμε την εξής ερώτηση. Αν ε, μια εμβάθυνση της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ε, θα κινδύνευε να μας βάλει σε μια πολύπλοκη κατάσταση απέναντι σε άλλους εταίρους, όπως η Ρωσία ή η Κίνα. Ξέρουμε ότι σε άλλες συμφωνίες, όπως με την Ουκρανία, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν ε, ίσως ποια είναι η κατάσταση και ποιο είναι ο αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συμφωνία στο επίπεδο αυτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Μιλάμε πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ μπόρεσα να εργαστώ στο πρωτόκολλο της Συμφωνίας για το Σμπεκιστάν και εργαστήκαμε πολύ με το Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας. Όμως, ε, ε, έχουμε ε, ουσιαστικά κάποιους δείκτες ε, του ΔΟΕ που είχε συνεργαστεί με τις αρχές του Ουσμπικιστάν. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε αξιολογήσεις και δείκτες που να μας επιτρέπουν να πούμε ότι γίνεται πρόοδος και υπάρχει θετική εξέλιξη ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι το Καζακστάν δεν είναι και μεγάλη δημοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Το τρίτο ερώτημα που θέτω για τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Το Καζακστάν ξεκίνησε μια διαδικασία με τον ΩΣΑ για να μπει ε, στην οικονομία της αγοράς. Εργαζόμαστε πολύ στο θέμα της οικονομίας της αγοράς. Έχουμε επίσης ενδείξεις ε, για την ε, εξέλιξη του ως προς ε, το αν προχωρά προς το να γίνει μια οικονομία της αγοράς και τις εργασίες που επιτελεί σήμερα με τον ΟΣΑ. Και το τελευταίο σημείο αφορά το συνδικαλιστικό ζήτημα. Μας έκρουσαν τον κόνδυνο του κινδύνου για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στο Καζακστάν. Πολλοί είναι φυλακισμένοι, απειλείται η συνδικαλιστική ελευθερία. Έτσι λοιπόν να προχωρήσουμε με μια χώρα που ενίοτε δείχνει να οπισθοδρομεί στο σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα ήταν ένα καλό μήνυμα να δώσουμε. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε πράγματι να έχουμε τους σωστούς δείκτες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω ε, άλλα αιτήματα για το, να πάρει το λόγο, ούτε άλλους και όδους εισηγητές. Λοιπόν, ερωτήσεις η Κομισιόν να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ερωτήματα. Πρώτον, η συμφωνία αυτή συνήφθη ή μάλλον η πρώτη ερώτηση αφορούσε τις επιπτώσεις προς τρίτους Ρωσία Κίνα, ας πούμε. Όπως γνωρίζουμε, το Καζακστάν ε, συμμετέχει στην Οικονομική Ένωση της Ευρασίας που είναι τελωνιακή ένωση και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο όταν συνήφθη αυτή η συμφωνία λάβαμε υπόψη μας τις υποχρεώσεις που έχει το Καζακστάν στα πλαίσια αυτής της Ένωσης και επίσης το γεγονός ότι εδώ δεν πρόκειται για Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, γιατί δεν είναι συμφωνία απελευθέρωσης ε, δασμών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης αυτής και δεν μπορούν να τα διαπραγματευτούν χωριστά τα μέλη της. Επίσης λαμβάνεται πλήρως υπόψη η συμμετοχή του Καζακστάν στην ε, Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Το ίδιο ισχύει και με τη συμφωνία που πρόσφατα συνήφθη με την Αρμενία ε, λάβαμε πλήρως υπόψη μας τους περιορισμούς που υπάρχουν λόγω της συμμετοχής στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Όπως είπα, η συμφωνία, στην εισαγωγική μου ομιλία, η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και αυτό για μας είναι σημαντικό στοιχείο τη θέμενη αξίας σε σχέση με τις προηγούμενες ε, συμφωνίες είναι ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δεσμεύσεις εφαρμογής των διαφόρων συμβάσεων στις οποίες ε, συμμετέχει το Καζαχστάν είτε στο τομέα, στον κοινωνικό τομέα είτε και στον περιβαλλοντικό τομέα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό μια χώρα όπως το Καζακστάν να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Κατά την ε, υλοποίηση της συμφωνίας όλα αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Συμμετείχα στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου και στο τέλος Μαρτίου φέτος για την νέα αυτή συμφωνία και ακριβώς ένα από τα θέματα που ε, τέθη στην εμπορική αυτή επιτροπή ήταν το θέμα της, ε, του κλεισίματος διαφόρων ανεξάρτητων ενώσεων και της σύλληψης ε, κάποιων ηγετικών στελεχών τους. Ζητήσαμε με την ευκαιρία εκείνη ε, από το Καζακστάν να επιτρέψει την ελεύθερη ε, ε, δημιουργία αυτών των συνδικάτων και την λειτουργία τους χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια και με την ευκαιρία εκείνη οι αρχές της χώρας μας ενημέρωσαν ότι σκόπευαν για μία ακόμα φορά να αναθεωρήσουν το συνδικαλιστικό τους νόμο για να ε, συνάδουν με τους νόμους και τα διεθνή πρότυπα. Επίσης καλέσαμε το Καζακστάν να απελευθερώσει τους ε, ηγέτες των τοπικών συνδικάτων Κουτσακ Μπάιεφ και Γελουσίνοφ που συνελήφθησαν και να σταματήσουν οποιαδήποτε κατασταλτικά μέτρα. Αυτά στα πλαίσια της ε, Επιτροπής ε, για τη Συμφωνία αυτή και της ευρύτερης ε, συμφωνίας που έγινε τις ημέρες εκείνες. Οπότε βλέπετε ότι στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας έχουμε περιλάβει και άλλα στοιχεία και επίσης συγκεκριμένους χώρους που, όπου ε, είμαστε σε θέση να θέσουμε επιτακτικά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα στο Καζακστάν. Και όσον αφορά την εργασία σε επίπεδο όσα, όπως γνωρίζετε το Καζακστάν δεν είναι μέλος του ΩΣΑ, όμως σκοπεύει να γίνει. Υπάρχει συνεργασία με τη γραμματεία του ΩΣΑ, την οποία παρακολουθούμε και η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Και άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα συζητηθεί την 30 Αυγούστου και ε, ελπίζω ότι θα υπάρχει και η τελική γνωμοδότηση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημεία 6 και 7. Ε, και φτάνουμε στο σημείο 8, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για τη στρατηγική ε, για το ε, ψηφιακό εμπόριο και θα δώσω μέσα τον λόγο στη συνάδελφο Μαρίκη και Σάκ. Χαίρομαι, λέει η κυρία Σάκε, γιατί έχουμε πλέον την ευκαιρία να συζητήσουμε επισήμως ε, την, ε, το έγγραφο εργασίας, ε, επί του οποίου παρακαλώ να συμβάλλετε έτσι ώστε να, γίνεται όσο, να γίνει όσο γίνεται πληρέστερη αυτή η εργασία ίδιας πρωτοβουλίας όσον αφορά το ψηφιακό εμπόριο και τη στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο. πιστεύουμε ότι ε, πρόκειται για μια σημαντική στρατηγική η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της

το διαρκώς και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αυτού του εμπορίου. Ε, η ψηφιακή επανάσταση έχει ε, ε, κατά πολύ επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων και φυσικά και την οικονομία γιατί ας πούμε ένας αρχιτέκτονας μπορεί πατώντας απλά ένα κουμπί να φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου στον πελάτη του. Θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη όλα τα επαγγέλματα γιατί ε, ξέρουμε ότι η ψηφιοποίηση αφορά πλέον όλους τους τομείς και όλες τους τομείς παραγωγής. Ε, είτε πρόκειται για παραγωγή προϊόντων, είτε υπηρεσιών, είτε πρόκειται για μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ε, δημιουργούνται και νέες ευκαιρίες μαζί με τις ε, γρήγορες ε, αλλαγές ε, και επομένως οι υφιστάμενοι κανόνες πλέον δεν αρκούν. Δεν έχουμε αρκετούς διεθνείς κανόνες και βλέπουμε ότι και οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου δεν κινούνται αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να έρονται τα εμπόδια τα οποία δημιουργούνται στην οικονομία. Μία τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ε, βλέπουμε ε, ε, εσωτερικές νομοθεσίες οι οποίες διαμορφώνουν την οικονομία και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να δούμε και τη διεθνή διάσταση αυτών των ε, κανόνων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ε, καλύτερη, ε, καλύτερη, δημιουργούν καλύτερες διαδικασίες. Ας πούμε υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδρυτής της Alibaba, Jack Ma, προωθεί τώρα μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παγκόσμιου εμπορίου ε, με την οποία επιδιώκει να δημιουργήσει εικονικές ζώνες ελεύθερου εμπορίου, οι οποίες θα επιτρέπουν στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ελεύθερα διασυνολογικές συναλλαγές χωρίς δασμούς. Αν δεν κινηθούμε γρήγορα λοιπόν, θα μας ξεπεράσουν αυτές οι καταστάσεις. Ε, θα πρέπει επομένως να προχωρήσουμε προς αυτό τον την κατεύθυνση, αλλά με τα απαραίτητα εχέγγυα και τους απαραίτητους και την τήρηση των απαραίτητων αξιών. Αυτές είναι οι αξίες, οι αξίες ευρωπαϊκή Ένωσης ε, θα πρέπει να διέπουν και αυτήν την ε, νέα στρατηγική. Ε, σωστή και δίκαιη πρόσβαση στην αγορά, διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων, παραγωγή αυτών ωφελών για τους καταναλωτές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό. Επίση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν, ας πούμε, να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το ψηφιακό εμπόριο ε, μέσω της διευκόλυνση, ας πούμε, της ψηφιακής ε, ε, υπογραφής, αλλά πάντα με σεβασμό των δικαιωμάτων και των καταναλωτών και την προστασία τους. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι ροέ των δεδομένων κάθε επιχείρηση η οποία ε, ασχολείται είτε με τα, τις υπηρεσίες είτε με τα προϊόντα ήδη ε, έχει ε, δεδομένα. Η δυνατότητα λοιπόν που θα έχει η κάθε επιχείρηση να έχει ελεύθερη ροή δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για το διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει επομένως να ε, λυθεί το ζήτημα αυτό οπωσδήποτε. Αυτό θα πρέπει να γίνει πάντα ε, με προστασία των ε, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Είναι, είναι λίγο ασαφή τα όρια ανάμεσα στον προστατευτισμό και την προστασία εντός ενός ελευθέρου εμπορίου. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Επίσης, να σας πω ότι ήδη από το 1998 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τηρείται ένα μορατόριο όσον αφορά τους δασμούς για τις ηλεκτρονικές ε, μεταδόσεις. Το, το μορατόριο όμως δεν αποτελεί μόνιμο μέτρο και επομένως υπάρχει κίνδυνος αύξησης των παγκοσμιών δεδομένων ε, που μπορεί να αποτελέσει ελκυστικό μέσο για δημιουργία εσόδων για τις ε, κυβερνήσεις. Ε, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα, στο οποίο θα ήθελα να με βοηθήσετε είναι η υποχρεωτική κοινοποίηση του πηγαίου κώδικα, η παράδοση των κλειδιών κρυπτογράφησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στην αγορά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι, σε ορισμένε χώρε ότι θα κοινοποιούν και θα παραδίνουν στο κράτο τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλων προϊόντων. Ε, υπάρχουν ε, τώρα νέες τεχνολογίες ε, κρυπτογραφήσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προϊόντα και χωρίς καμία μείωση της κυβερνόπροστασίας. Επίσης θα πρέπει να δούμε και στοιχεία που αφορούν ας πούμε την ασφάλεια, τα διεθνή πρότυπα ε, συγκεκριμένη διατύπωση όσον αφορά την ε, προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων. Βεβαίως, ε, η γνωσιοκεντρική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ ψηλά στην αλυσίδα αξίας, αλλά είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε μια νέα ισορροπία. Έχουμε μάθει ε, ε, με την όκτα ας πούμε, μαθήματα από το παρελθόν και επομένως τα ψηφιακά δικαιώματα ε, είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να, να ξεκαθαρίσουμε τι θα πρέπει να καλύπτεται και να προστατεύεται ως διανοητικό δικαίωμα και τι όχι. Τέλος. Κυρίως όσον αφορά τις ε, ε, υπηρεσίες, ε, η πρόσβαση στην ψηφιακή υποδομή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρχει η πρόσβαση απαραίτητη ε, στην ψηφιακή ε, υποδομή ε, και κυρίως η πρόσβαση στα δίκτυα τρίτων χωρών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη στρατηγική προς την ψηφιακή αγορά. Τέλος, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε εδώ μόνο με όρους προστασίας της αγοράς αλλά και προστασίας των ανθρώπων θα πρέπει να δούμε με, κατά πόσον μπορεί μια τέτοια εμπορική ψηφιακή πολιτική και μια πολιτική ψηφιακού ε, εμπορίου να βοηθήσει ή στην υλοποίηση των βιώσιμων στόχων ε, ανάπτυξης, ε, ας πούμε ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, επιγραμμικών ε, ικανοτήτων για ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα αυτές τις δυνατότητες. Επίσης το θέμα της ουδετερότητας του δικτύου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μαζί με άλλα στοιχεία εξίσου σημαντικά όπως η κρυπτογράφηση ας πούμε με ταυτόχρονη προστασία βεβαίως της ελευθερίας του λόγου των ανθρώπων κλπ αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να σας πω, ε, ε, να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν ε, κατά κάποιο τρόπο τον κορμό της εργασίας μου. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη τροφή προς σκέψη και θέλω και την βοήθειά σας, το input σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο πλήρη εργασία. Είμαι εδώ, είμαι ανοιχτή στις ιδέες σας, είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, αυτή η έκθεση και κυρίω σε ό,τι αφορά και τη συζήτηση στο ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και στα πλαίσια της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας αυτή η συζήτηση για τη ρύθμιση της ροή των δεδομένων και της προστασίας των πιστωτών. Θα δώσω τώρα το λόγο στους και εισηγητές για το ΕΛΚ. Ο κύριος Βαλές από την Βιάν Ρέντινγκ. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντινγκ μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή τη. Ε, συμφωνεί με την άποψη ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό γραφό εργασία ε, που καλύπτει όλα τα στοιχεία σχεδόν, τα οποία αναφερόμαστε συνήθως ως ψηφιακό εμπόριο. Κάνει τη σωστή διάκριση μεταξύ του θα πρέπει να συμπεριληφθεί στι εμπορικέ συμφωνίε, παραδείγματο χάρη ένα μορατόριο για του δεσμού για τι ηλεκτρονικέ μεταδόσει και η μεγαλύτερη πρόσβαση στι αγορέ τηλεπικοινωνιών και τι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, παραδείγματο χάρη προστασία των δεδομένων και το copyright. Η κυρία Ρέντινγκ επίση συμφωνεί με το στόχο Τη εισηγήτρια ε, να τροποποιηθούν οι διεθνείς κανόνες για να προστατευτούν καλύτερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και να υποστηριχθούν καλύτερα οι ευρωπαϊκές εταιρείε. Ε, θα είναι πολύ σημαντικό το έργο μας, το φάκελο αυτό, εν ώψη της Υπουργικής του ΠΟΕ που θα λάβει η χώρα στον πένο στο στο Δεκέμβριο, όπου το ψηφιακό εμπόριο βρίσκεται στην κορφή τη ημερησία διάταξη. Αυτά προετοιμάσει η κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και η Καρολίνα για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πολύ ισορροπημένο κείμενο που έχουμε. Καλύπτει πολλούς τομείς και μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία. Βέβαια, πιστεύουμε ότι λείπουν ένα-δύο πράγματα. Προφανώ ε, θα πρέπει να είναι καλά διαρθρωμένο το ψηφιακό εμπόριο, γιατί αποτελεί το μέλλον και θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ποιο το μισκαλύπτει. Αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εμπόδια εμπορικά σε πολλούς τομείς. Την ε, πρώτη φορά που το συζητήσαμε αυτό, είπαμε ότι πρέπει να βρούμε και τη μέση εδώ μεταξύ του προστατευτισμού και του υπερβολικού φιλελευθερισμού στην έκθεση αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ε, μία ισορροπία μεταξύ απόλυτα ελεύθερη ροή ε, δεδομένων και τη αποθήκευση των δεδομένων από την άλλη. Ούτε θα πρέπει να ξεχνάμε την προστασία των δεδομένων. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλά τα πρότυπα στην Ευρώπη για την προστασία των δεδομένων και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα σεβόμαστε αυτά. Φυσικά θέλουμε να διατηρήσουμε το ανοιχτό ίντερνετ και να διατηρήσουμε την ελεύθερη ροή των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε τα spam, να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή και να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Επίσης, ε, θα πρέπει να εμποδίσουμε το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων ε, μέσω του εντοπισμού. Χρειαζόμαστε μια ψηφική στρατηγική που να δίνει ασφάλεια και να μπορεί να εγγυηθεί την προστασία του ιδιωτικού χρήστη, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί ένα ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο και δημιουργεί και ανταγωνισμό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε εμπόριο για όλους. Κατόπιν έχουμε και τους δασμούς τους τελωνιακού δεσμούς ε, και το χάρη μπορούν να υπάρχουν δασμοί ε, όπως ε, στα ηλεκτρονικά βιβλία, στη μουσική και σε άλλα αγαθά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα της απλούστευσης του εμπορίου και θα πρέπει να έχουμε και ευφύς συναλλαγές χωρίς έγγραφα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα δικαιώματα του καταναλωτή. Η προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ε, ότι όταν ε, αγοράζουν ε, υπηρεσίες πληρούνται και τα κατάλληλα δεδομένα, τα δικαιώματά τους ε, προστατεύονται και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, να δούμε και πτυχές όπως ε, η ευθύνη στο διαδίκτυο και τι γίνεται με τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και τις νοσίστατες επιχειρήσεις, τις startup. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική και για αυτές. Πρέπει να μπορούμε να ανταγωνιστούμε, αλλά χρειαζόμαστε κανόνες που να μπορούν να γίνουν σεβαστοί από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο από τις μεγάλες εταιρείες ή τις πολυεθνικές η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι δομές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να επενδύσουμε στην υποδομή γιατί έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Οι αναπτυσσόμενες χώρες επίσης έχουν ευκαιρίες και είναι ανταγωνιστικές. Και κάτι τελευταίο για μένα σημαντικό είναι το εξής οι νέες ε, πλατφόρμες, ε, ψηφιακές πλατφόρμες και ψηφιακοί χώροι εργασίας. Θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε αυτό σαν crowd working. Αυτό ε, ουσιαστικά διέπεται από ένα περιβάλλον που είναι φορτωμένο με υπερβολικούς κανόνες. Αυτές οι δουλειές θα πρέπει να είναι ασφαλείς, καλές δουλειές και ξέρω ότι ακόμη και αν δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας είναι ένα θέμα που θέλω να θίξω γιατί ξέρουμε ότι αυτού του είδους οι θέσεις εργασίας αυξάνονται. Χρειαζόμαστε δίκαιο ψηφιακό εμπόριο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μπορούν όλοι να συμμετέχουν και όλοι να υποφεληθούν από αυτό. Ανυπομονώ να δω το σχέδιο της έκθεσης και ανυπομονώ να συνεργαστώ και με την εισηγήτρια τις επόμενες ημέρες για να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ λέει ο κύριο Σόλτ. Ε, κοιτάξτε, έχουμε αλλάξει τι αρμοδιότητε στην ομάδα μα. Εγώ έχω αναλάβει το φάκελο και θέλω να ευχαριστήσω σήμερα την κυρία Σάκε που μα ε, παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο εργασία. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση και έχουμε ε, ουσιαστικά πολλές προκλήσεις για το μέλλον του διεθνούς εμπορίου. Όλοι γνωρίζετε πώς ε, το διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση αλλάζουν τις οικονομικές εξελίξεις. Και φυσικά επηρεάζουν και το εμπόριο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλες χώρες. Ε, στην ψηφιακή εποχή, η ψηφιοποίηση της οικονομίας νομίζω θα μπορούσε να είναι η ψηφιοποίηση της οικονομίας μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Και επομένως ένα ρυθμιστικό πλαίσιο χρειάζεται. Και φυσικά και στην αρχιτεκτονική για το διεθνέ εμπόριο. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου ε, έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές, το διαδίκτυο επιτρέπει στις επιχειρήσεις ε, να συμμετέχουν. Το διαδίκτυο έχει γίνει σημαντικό εργαλείο για τι επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με του καταναλωτέ και του προμηθευτέ, ε, για ε, να έχουν χρηματοδότηση από το είναι πληθωριστική χρηματοδότηση, ε, να διαχειρίζονται διάφορα προϊόντα, να συνεργάζονται με τοπικούς ερευνητέ κτλ. Όλε αυτέ οι δραστηριότητε μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένε ευκαιρίε και για του καταναλωτέ και για του παραγωγού μέσω του διεθνού εμπορίου. Ταυτόχρονα όμω, Όλες αυτές οι πτυχές ε, ανοίγουν, ε, ε, ανοίγουν νέα ζητήματα για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων, την ιδιωτική σφαίρα κτλ. Η συγγήτρια ήδη προσπαθεί να επικεντρωθεί στη μία ή στην άλλη πτυχή. Συμφωνώ ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να δημιουργήσει αυτά ωφέλη για τους καταναλωτές και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός θα πρέπει να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων ε, και να πετύχει παγκόσμια γνώση. Επίσης, θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μας στο εξή. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα πιο σαφή χαρακτηρισμό για το τι πράγμα μιλάμε όταν αναφερόμαστε στο ψηφιακό εμπόριο. Το ψηφιακό εμπόριο θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στη βιομηχανική πολιτική, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα ιδιωτικό ζήτημα και συμφέρον. Ε, ουσιαστικά ε, ενδιαφέρει και τις διάφορες ε, βιομηχανίες. Έχουμε διάφορες πτυχές μέσω της παραγωγής, μέσω της κατανάλωσης και μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να θίξω και άλλε δύο πτυχέ. Τα μαζικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτική ζωής. Άκουσα και το σχολείο της κυρίας Ρέντινγκ, συμφωνώ. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες. Όμως θα πρέπει να είναι σαφές ότι και οι πολίτες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής και τα δεδομένων. Θα έχετε διαβάσει τι ε, συμβαίνει με τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται η κυβέρνηση, που διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις. Ουσιαστικά θα πρέπει εμείς να τονίσουμε το θέμα της προστασίας των δεδομένων και να το διασφαλίσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν αποτελούν εμπόδιο στο εμπόριο, αλλά θα θεμελιώδη δικαιωμένα οι ροές των δεδομένων αφορούν και ροές προσωπικών δεδομένων. Και θέλω να επιστήσω την προσοχή μας ε, στην υπουργική δήλωση που προέκυψε από τη συνάντηση στο ΩΣΑ πρόκειται για ένα τεράστιο έγγραφο και αναφέρονται πάρα πολύ σε αυτή την πτυχή της ανταλλαγής των δεδομένων προς το συμφέρον των ανθρώπων, αλλά φυσικά δημιουργούνται και ευκαιρίες για κατάχρηση των δεδομένων. Παραδείγματο χάρη, οι χώρες που διαπραγματεύονται με τις, την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Δεν είναι η νομοθεσία τους απαραίτητα στο επίπεδο που αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, τι δεσμεύσει θα αναλάβουμε σε ό,τι αφορά την ελευθερία, την ελεύθερη ροή των ε, δεδομένων. Χρειαζόμαστε ένα σαφή ορισμό εδώ. Τώρα, το άλλο θέμα είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουμε έναν επιστήμονα από την ε, Γερμανία, Hans Beckler, ο Τζικριτής ε, αναλύει ότι μέσω της ε, οικονομίας του επιμερισμού υπάρχουν νέες οικονομικές εξελίξεις. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σήμερα. αλλά θα ενημερώσω την εισηγήτρια και τους και τους εισηγητές για τα θέματα αυτά. Τώρα, ε, για την ε, μερισμένη οικονομία. Νομίζω ότι δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ε, και ευελιξία, αλλά η ευελιξία πολλές φορές σημαίνει επισφάλεια δεν ε, μπορούμε ε, να αγνοήσουμε ότι εμφανίζεται ένα νέο είδος επισφάλειας, επισφαλή επισφαλής εργαζόμενη. εργαζόμενη. Οι άνθρωποι που είναι αυτοπασχολούμενοι στον ε, ψηφιακό τομέα χρειάζονται προστασία οι χειριστές ε, των πλατφορμών online θα πρέπει να θέσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να διαπραγματευτούν συλλογικά για αξιοπρεπείς μισθούς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς κανόνες ε, και να αποφύγουμε οι πλατφόρμες να γίνουν παράδειση φοροδιαφυγής και αποφυγής καταβολής ε, των κοινωνικών εισφορών. Πιστεύω ότι η ψηφική οικονομία μας ε, επιτρέπει ψηλά ε, κινητή κατανομή ε, των διάφορων καθηκόντων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μοντέλα επιχειρηματικά διαφορετικά. Εδώ η εμπορική πτυχή της ψηφιοποίησης της οικονομίας συνδέεται άμεσα και στις ικανότητες των κοινωνιών μας να φορολογήσουν ε, τα άτομα και θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία επιβεβαίωσε ότι η ψηφιοποίηση παίζει έναν θεμελιώδη ρόλο για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο διαδίκτυο και 90% από αυτού βρίσκονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα είναι πολύ σημαντικό για να έχουν όλοι ίση πρόσβαση στη γνώση και στην ενημέρωση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει με τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ. Κύριε Ο κύριο Μπίτικοφ είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ την εισηγήτρια για ένα πολύ εύληπτο και σαφές έγγραφο εργασίας. Τώρα, μόνο ε, κάνοντας δύο ερωτήσεις μπορώ να συνεισφέρω στη συζήτηση. Πρώτον, το έγγραφο εργασίας θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πρότυπα. Εμείς πιστεύω ότι παρακολουθούμε έναν αγώνα θέσεως προτύπων ή ρυθμιστικών, ε, ένα ρυθμιστικό αγώνα. Και το αναφέρει αυτό κατά κάποιο τρόπο και η συγγήτρια όταν παίρνει παραδείγματα από τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα στην, ε, στο κείμενό της. Αν επικεντρωθούμε στην εμπορική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην ε, την πολιτική του εμπορίου και αυτό αναφέρεται και στις γενικές αρχές. Πρώτον, η εξασφάλιση της ε, δίκαιης πρόσβασης στην αγορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις τρίτες χώρες. Φυσικά είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ο τρόπος με τον οποίο, σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα ε, μεταφερθεί στην πράξη, πώς θα ερμηνευτεί αυτό στην πράξη. Η συγγήτρια χρησιμοποίησε και αλλού στο κείμενο τον όρο αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά. Εδώ όμως η αμοιβαιότητα δεν αναφέρεται ρητά. Θα πρέπει αυτό να αποτελέσει ένα μια πολιτική αρχή που θα την συμπεριλάβουμε όταν ε, ε, μιλάμε για δίκαιη πρόσβαση στην αγορά τις διάφορες πολιτικές με βάση τις οποίες η χώρα, οι χώρες θα επιμένουν στο θέμα του εντοπισμού των, data localization ή που θα το απορρίπτουν ή τις ε, απαιτήσει αποκαλύψεων που επίσης, με τις οποίες επίσης δεν συμφωνούμε. Η πολιτική ψηφιακού εμπορίου που πρέπει να ακολουθήσουμε ποια θα είναι. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω αφορά τη ροή των δεδομένων. Θέλω κάποιες, κάποια διευκρίνηση από την εισηγήτρια. Θεωρείτε ότι ότι οι διαμεθοριακές ροές δεδομένων είναι ο τρόπος το, για να επιτευχθεί αυτό το advocacy επίσης θεωρείται ότι ε, οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την ρυθμιστική σύγκληση στο τομέα του ψηφιακού εμπορίου ή θεωρείται ότι αυτού του είδους η συνεργασία θα πρέπει να επέλθει σε άλλα ειδικά για αυτό το σκοπό ε, ε, διεθνή φόρα. Και τέλος, όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα, θεωρώ η τυποποίηση είναι μέρος του όλου αυτού ανταγωνισμού για τα θεσμικά, για τα ρυθμιστικά θέματα και ότι τα, οι διεθνείς οργανισμοί που θέτουν τα πρότυπα δεν έχουν πάντα τον έλεγχο της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, παρότι είμαι υπέρ της συνολικής στάσης του εγγράφου εργασίας δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτούς τους οργανισμούς που θέτουν τα διεθνή πρότυπα και διαρωτώ αν όντως μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο που αναμένεται από αυτούς να παίξουν. Ευχαριστώ. πολύ. Αλλά και εγώ έχω σκεφτεί αυτό το θέμα της, ε, των ροών δεδομένων. Υπάρχει η ανάγκη, όπως γνωρίζετε, να συζητηθεί λεπτομερέστερα το θέμα. Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε ροή δεδομένων σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Έχουμε το 14 συν του ΓΚΑΤΣ. Είναι αυτός ο τρόπος που θα μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε. Πιστεύω ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή θα κινηθεί προς το να πει ναι, αυτό είναι, αυτή είναι η κατεύθυνση, να γίνει πλήρης εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων και να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση των ε, συστημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και μετά να προχωρήσουμε στις ροές δεδομένων. Αυτό θέλετε να συμβεί στη διαπραγμάτευση της προστασίας των δεδομένων σε κάθε ε, συμφωνία ελευθερών εμπορίου, γιατί με την Ιαπωνία το επίπεδο είναι λίγο πολύ παρόμοιο. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην αμοιβαία αναγνώριση, αλλά υπάρχουν και χώρες όπου το επίπεδο προστασίας δεδομένων είναι χαμηλότερο. Ίσως η Κομισιόν να το σκεφτεί αυτό και τα άλλα ερωτήματα που ανέφερε η συγγήτρια και οι σκιώδες εισηγητές. Και ο, ο Κρίστοφ Κίνε θα απαντήσει εκ μέρους της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και όπως και οι άλλοι ομιλητές να ευχαριστήσω την κυρία Σάκε για την φιλόδοξη ε, και πολύ ε, συνολική προσέγγιση που έχει ακολουθήσει ε, σε αυτό το έγγραφο παρότι το θέμα είναι πολύ τεχνικό. Θα ήθελα να πω ότι για θα θέλαμε να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα ευμενές περιβάλλον για την ψηφιοποίηση, την πρόσβαση στην αγορά ε, και η προστασία των καταναλωτών και η δικαιοσύνη βεβαίως αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας. Βεβαίως προσπαθούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουμε αυτό που θέλουμε ε, και θέλουμε και μια προσέγγιση ελευθέρου εμπορίου που σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο κεφάλαιο ε, στη, για την ψηφιοποίηση στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, παράδειγμα ας πούμε το, η πρόσφατη συμφωνία με την Ιαπωνία και ε, ε, μάλιστα μπορώ να σας πω ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα από τα στοιχεία που ακούσαμε, περιλαμβάνονται στη συμφωνία με την Ιαπωνία. Επίσης θα θέλαμε ε, να είμαστε ε, να, να προωθήσουμε ένα τέτοιο θέμα και ένα αντίστοιχο θεματολόγιο στην, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά ο αριθμός των χωρών είναι τέτοιος ε, που ε, ε, μοιραία και μηχανικά το όριο της φιλοδοξίας σίγουρα χαμηλώνει. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι και πρόσφατα στην Γενέβη τις τελευταίες εβδομάδες υπεραμείνθηκα προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πρόβλημα να πείσουμε κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες για την αξία της ψηφιοποίηση. Ε, όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά, το στήμα 3 ας πούμε της ε, εκθέσεως ε, και αναφερόμενο στο 3.1 ροές δεδομένων, πιστεύω ότι είναι σαφής η ανάγκη να εξευρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην αφενός προώθηση ενός ε, ε, φιλόδοξου θεματολογίου ε, που θα αφορά τις ροές δεδομένων, τις τις πρακτικές για την τοπικοποίηση δεδομένων κλπ. από τη μία πλευρά και την γενικότερη ισορροπία του εμπορίου από την άλλη. Εμείς πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε αυτήν την ισορροπία. Η Κομισιόν συγκεκριμένα προσπαθεί να βρει καλή διατύπωση η οποία θα μπορέσει να ε, συνδυάσει τους δύο στόχους και θα διασφαλίσει ότι και οι δύο πυλώνες μπορούν να προχωρήσουν ε, με αμοιβαία υποστήριξη. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει και ε, διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο για το Concept Paper, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Ενδεχομένως ε, βεβαίως θα πρέπει και να ε, πάρουμε διδάγματα από την πρόσφατη συμφωνία και τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Ε, ίσως μια ιδέα για το έγγραφο εργασίας θα ήταν να αναφερθεί και στον δυνητικά καλό ρόλο που σχετικές αποφάσεις συμμόρφωσης For uh, ε, μπορούν να παίξουν στον ε, τομέα αυτό. και βεβαίως πάντα με, ε, στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στη συμφωνία με την Ιαπωνία είχαμε την δήλωση των προέδρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφενός και του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας κατά την έννοια αυτή. Επίσης, Υποστηρίζουμε τα στοιχεία για τους ε, δασμούς στις ηλεκτρονικές ε, ε, μεταδόσεις όσον αφορά το μορατόριο και επίσης την υποχρεωτική κοινοποίηση του πηγαίου κώδικα ή την παράδοση των κλειδιών κρυπτογράφησης. όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα για τα ψηφιακά προϊόντα, ναι, και με αυτό συμφωνούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Ε, γιατί όντως ε, δεν ορίζονται τα πρότυπα από τις συμφωνίες ε, εμπορίου. Για την διανοητική ιδιοκτησία μπορούμε να συμφωνήσουμε με το κείμενο έτσι όπως έχει διατυπωθεί. Πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές εδώ. Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές ε, ε, επιχειρήσεις επικοινωνία έχουν και θα έχουν πρόσβαση στην τοπική αγορά. Αυτά και από οικονομικής και από άλλες απόψεις είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ε, επίσης ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε και με την ε, επιθυμία που εκφράστηκε, την ευχή που εκφράστηκε για την περιαγωγή. Βέβαια νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν μέσω της συμφωνίας των εμπορικών συμφωνιών, είναι υπερβολικό να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίτευγμα το απίστευτο που είχαμε όσον αφορά την περιαγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Να πω και δύο λόγια σχετικά ε, με τη, το με τη στρατηγική ψηφιακού εμπορίου ε, που θα βασίζεται σε αρχές ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε και από πλευράς της Κομισιόν ότι αυτό είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό και επομένω, η Κομισιόν μπορεί να συμφωνήσει με την στρατηγική έτσι όπω αναφέρεται στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μαρία Διεσάκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τόσο μεγάλο κατάλογο προτάσεων, σχολείων, σκέψεων. Νομίζω ότι αποτελεί μια καλή βάση να εργαστούμε περαιτέρα και να αποσαφηνίσουμε για το τι πράγμα μιλάμε. Θα κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με το τι θα έπρεπε να είναι εντός και τι θα έπρεπε να είναι εκτός ε, οποιασδήποτε εμπορική συμφωνίας όταν μιλάμε για τις ροές δεδομένων. Δεν ε, μπορώ παρά να τονίσω καταρχήν ότι πρέπει να εργαστούμε βάσει αρχών που δεν είναι επίμαχες και που περασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουμε τρόπους για το πώς μπορούμε να τις εντάξουμε στις εμπορικές συμφωνίες. Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει δυνατότητα ε, να βάλουμε τους ε, κανόνες για τις ώρες δεδομένων, δεν είναι οι εμπορικές συμφωνίες το σημείο που πρέπει να αναφερθούμε στην προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων ή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ουσιαστικά ε, μέσω των ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων δεν αλλάζουμε το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα που αναδύονται στις συζητήσεις μας και νομίζω ότι και εδώ είναι σχετικό. Τώρα θα σας δώσω όμως ένα παράδειγμα της ιδέας των προτύπων και για να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Μπουτικόφερ. Αν δείτε το δίκτυο των πραγμάτων, της εφήσεις συσκευές, ήδη ε, κυκλοφορούν στην αγορά αυτές οι εφήσεις συσκευές και ε, ε, γίνονται εισαγωγές σε όλο τον κόσμο, χωρίς διεθνείς κανόνες για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο μη ασφαλών συσκευών που θα έχουν αντίκτυπο και στην ιδιωτική ζωή και στα δεδομένα, στην ασφάλεια των δεδομένων των ανθρώπων, αλλά και στην ασφάλεια των δικτύων. Επομένως, βλέπουμε ήδη ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει τώρα να έχουμε κανόνες και να ελεγχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο στην περίπτωση του δίκτυου των πραγμάτων. Το ψηφιακό εμπόριο δηλαμβάνει χώρα και το εμπόριο στα ψηφιακά αγαθά ή χώρα και δεν έχουμε κανόνες. Και οι κανόνες καθυστερούς χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πολιτικό όραμα τεχνικής κατανόησης για το τι είναι ήδη δυνατόν ε, και για το πού μπορεί να μας οδηγήσουν οι μελλοντικέ εξέλιξεις ε, και κατόπιν βάση αυτού του πολιτικού οράματος ε, να έχουμε ένα σύνολο αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από αυτό το όραμα μπορούμε σε κάθε συμφωνία, σε κάθε απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί, μπορούμε να εξετάζουμε ποιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι απαραίτητες όχι μόνο από τη δική μας κοπιά των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών εταιριών, αλλά να έχουμε και αυτή την παγκοσμία ευθύνη για το τι μπορούμε να πετύχουμε στις τρίτες χώρες, όπου συχνά δεν έχουν αναπτυχθεί πρότυπα ή κανονισμοί. Και υπάρχει και η πολιτική ευκαιρία. Το είδαμε ήδη αυτό. Πολλέ φορέ στρέφονται οι αναπτυσσόμενε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταφέρουν στο δικό του δίκαιο κάποιου από του κανόνε και την ομοθεσία που έχουμε αναπτύξει εδώ. Θέλουν να πετύχουν λοιπόν παρόμοια πρότυπα και να διευκολύνουν και την πρόσβαση στην αγορά. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε ακριβεί και να καταλάβουμε τι τεχνικέ πραγματικότητε. Έτσι μπορούμε να εργαστούμε περαιτέρω. Είναι σημαντικό να έχει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η ζωή ενώ εμείς αναπτύσσουμε αυτή τη στρατηγική και ίσως ε, θα μπορούσαμε να είμαστε σε έναν ε, αγώνα ε, στον υπόδρομο, όπως είπε ο κύριος Μπουτικόφορ. Δεν θέλω να μιλήσω για έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω, τα πρότυπα που τίθεται σε ιδιωτικό επίπεδο είναι μία εντελώ μια διάσταση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί γιατί εμεί θα πρέπει να λειτουργήσουμε έχοντας κατά νου το δημόσιο όφελος. Θα σταματήσω εδώ. Σημείωσα όλες τις ερωτήσεις και τις προτάσεις. Φυσικά αυτό ήταν ένα σχέδιο του εγγράφου εργασίας, θα ακολουθήσει ένα σχέδιο έκθεσης και κατόπιν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα περαιτέρω στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ Μαρίκη. Πράγματι ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με βάση του εγγράφου αυτού και περιμένουμε το σχέδιο έκθεση 25 Σεπτεμβρίου, οπότε θα γίνει συζήτηση επί της έκθεσης για μια ακόμη φορά και σε 9 Νοεμβρίου θα, θα υποβληθούν οι ε, τροπολογίες και το Νοέμβριο θα γίνει η ψήφιση εν ώψη του Buenos Aires, της Υπουργικής του Buenos Aires. Ευχαριστούμε πολύ στο σημείο αυτό. Ολοκληρώνεται η συζήτηση επί του θέματος 8 και τώρα περνάμε στο σημείο 9, το οποίο θα συζητηθεί in camera και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό το λόγο θα διακόψουμε για δύο λεπτά, τρία λεπτά θα επιτρέπεται να παραμείνουν μόνον όσοι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην αίθουσα.